δύο ε, συναδέλφων. Εξάλλου, έχει κατατεθεί αίτηση άρσης ασυλία του Μπόλου και η αίτηση αυτή με βάση το κανονισμό θα διαβιβαστεί στην ε, αρμόδια Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Θα ήθελα επίσης ε, να σας